Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. I welcome again to Brussels. <laughs> Καλώς ήρθατε και πάλι στις Βρυξέλλες μετά τις θερινές διακοπές. Ελπίζω να περάσατε καλά. Πραγματικά μου έλειψε αυτή η βροχή. Με το που έφτασα όμως στις Βρυξέλλες διαπίστωσα πόσο σημαντική είναι η βροχή στο Βέλγιο. Ας αρχίσουμε όμως με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Έχετε λάβει το σχέδιο. Αν σας κάνω κάποιες παρατηρήσεις, ο συνάδελφος Γιώργ Λάιχτφριντ, ο εισηγητής μας δηλαδή για μία από τις εκθέσεις που θα ψηφίζαμε κανονικά σήμερα, μου ζήτησε να αναβάλουμε τη συζήτηση για το σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης, την τροποποίηση του κανονισμού για την θέσπιση καθεστώτος, για την εξαγωγή κάποιων προϊόντων διπλής χρήσης και τεχνολογίας. Οπότε αναβάλλεται το σημείο 13 κατά έτσι του εισηγητού Γιώργ Λάιχτφριτ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ενημέρωσε ότι δεν θα παρεστεί στο σημείο 14 της σημερινής διάταξης. Το σημείο 14 προβλέπει συζήτηση της νέας ενεργειακής στρατηγικής για την Ευρώπη. Ο Γιάννης Σαχραντήλ δυστυχώς δεν θα μπορέσει να είναι εδώ. Ο κύριος Αρίφ ζήτησε το λόγο. Για το σημείο 12, κύριε Πρόεδρε, μήπως θα μπορούσαμε να αναβάλουμε τη συζήτηση. Γιατί πολλές ομάδες δεν έχουν ορίσει ακόμη τον εισηγητή του στο ίδιο και δική μου. Και θα προτιμούσα να αναβληθεί η συζήτηση αυτή για μετά το Στρασβούργο, ώστε να προλάβουν και οι ομάδε μεταξύ των άλλων και η δική μου πολιτική ομάδα, να ορίσουν του εισηγητέ του. Οπότε ζητήσατε να αναβληθεί το σημείο 12. Καλώς, θα το αφήσουμε για άλλη φορά. Οπότε αναβάλλεται και το 12 μαζί με το 13. Συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη όπως έχει τροποποιηθεί. Ωραία, εγκρίνεται λοιπόν. Σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών των δύο τελευταίων συνεδριάσεών μας του Ιουνίου και Ιουλίου. Αν δεν υποβληθούν σχόλια ή αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασής μας, θα θεωρηθούν συγκεκριμένα τα πρακτικά. Σημείο 3. Ανακοινώσεις ε, του Προέδρου. Η σύντηση της Επιτροπής μας αναμεταδίδεται απευθείας, εκτός από το τμήμα που θα γίνει και κλεισμένο το θηρό φυσικά. Και όλα τα έγγραφα έχουν διανεμηθεί. Και το σημείο 5 από το newsletter μόλις τώρα κυκλοφόρησε και ευχαριστώ θερμά τη γραμματεία για την καταπληκτική δουλειά της. Ας περάσουμε στις ψηφοφορίες τώρα. Σημείο 4. Prepare your voting card. Ετοιμάστε παρακαλώ τις ε, ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας. Το πρώτο σημείο είναι η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Εισηγητής ο Ιούλιο Βίνκλερ του ΕΛΚ. Έχουμε εξετάσει τις τροπολογίες στον Ιούλιο, τις 5, και από ό,τι ξέρω το Συμβούλιο συμφωνεί με τις τροπολογίες μας, οπότε μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία ήδη με την πρώτη ανάγνωση. Αλλά ας δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον Ιούλιο Βίγκλερ, για να μας πει αν έχει κάτι. Ευχαριστώ. Θα είμαι λακωνικός γιατί η συζήτηση ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο, όταν ψηφίσαμε και τις τροπολογίες. Θα ήθελα απλώς να ενημερώσω τους συνα... ότι οι τροπολογίες αυτές ξεκίνησαν από τη συζήτηση που είχαμε για την μακροοικονομική συνδρομή στην Ουκρανία, που και εμπνευστήκαμε τις τροπολογίε και για τη Μολδαβία. Θέλουμε διαφάνεια, έλεγχο τους, του Κοινοβουλίου και διάφορα άλλα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις τροπολογίε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Μολδαβία, γιατί βρίσκεται σε δινή οικονομική κατάσταση η χώρα αυτή, που είναι η γειτονική χώρα και περιμένει πώς και πώς αυτό το σημαντικό μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό καλύτερα να ψηφίσουμε το συντομότερο δυνατό. Ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Περισσεύει μία ψήφος πρασίνων. Παρακαλώ κάποιους από τους πράσινους να αφαιρέσει την κάρτα του από το μηχάνημα. Who, who, how many votes do they have? Two. Two. So who? Two votes. Οι πράσινοι δικαιούνται δύο ψήφους. αλλά κάποιος ψηφίζει χωρίς να το δικαιούται. ομόφωνη. Η Επιτροπή μας εγκρίνει το σχέδιο. Συγχαρητήρια. ψηφί. εγκρίνεται η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή προς τη Μολδαβία. Α, δεν είπατε τίποτα, έπρεπε να το είχατε δηλώσει. Ότι είχε πρόβλημα το μηχάνημά σας. Υπάρχει μία ψήφος κατά, άρα δεν ήταν παψήφη έγκριση. 20 υπέρ, μία ψήφος κατά. Τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος. Το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά δεν φαίνεται και πάλι αρνητική ψήφος. Ε, μετακινηθείτε για να ψηφίσετε σε άλλο μηχάνημα. Καλώς, το σημειώνουμε μία ψήφος κατά. Οπότε συγχαρητήρια. Τελειώσαμε με την ψηφοφορία στο 4. Σημείο 5. Τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου για τα εξαιρετικά μέτρα σε χώρες ε, που συμμετέχουν συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίηση και σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος είναι ο εισηγητής. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά πρώτα την τροπολογία 3. Ή μάλλον όχι, την έχω αποσύρει, λέει ο πρόεδρος. Η μαλλον οχι την εχω αποσυρει λεει ο προεδρος τροπολογια 4. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές. Οι υπόλοιποι υπέρ. Τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Μία αποχή. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με μία ψηφοκατά. Τροπολογία 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με μία αποχή. Τροπολογία 8, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται με μία ψηφο Τροπολογία 9, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται ομόφωνα. Τροπολογία 10, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται με μία ψηφο κατά, τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογικές και ψητιολογική έκθεση. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, με μία ψήφο κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με μία αποχή. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. για την πρόταση επιτροπής μας όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Βίλιαμ, ψηφίσετε κατά. Όχι, μεσαγυνεύσατε και ψήφισε υπέρ. Ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. εγκρίνεται με μία αποχή. Ψηφίζουμε την έναρξη άτυπων διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Ποιος είναι υπέρ για την σύναψη εγκαιρών συμφωνιών, αποχέ, ε, κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στο σημείο 6, θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο για όλα τα τμήματα. Ο Πέτερ Στιάστνη είναι ο εισηγητής μας από το ΕΛΚ. Let's start by the amendments on the draft Λοιπόν, να πιάσουμε πρώτα τις τροπολογίες στο σχέδιο γνώμης. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές αν δεν κάνω λάθος ελέγξαμε. Α, θα, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχιδη ψηφοφορία. ακολουθήσατε τη συμβουλή μου. Πέρα της ψηφοφορία, λοιπόν το αποτέλεσμα είναι ε, θετικό, όχι αρνητικό. Με συγχωρείτε όλοι, ο πρόεδρος ε, είναι αρνητικό, απορριπτικό. Όχι, λάθος, λάθος, λάθος. Κοιτούσα λάθος του αριθμούς. Αρχίζω με την παράγραφο 4, το αρχικό σχέδιο κειμένου, τμήματική ψηφοφορία, το πρώτο τμήμα. Α, όχι, όχι. Όχι, όχι. Καταπίπτουν τα δύο τμήματα και προχωρούμε στην παράγραφο 5 και στην τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Είναι η τροπολογία 8. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πάμε στη 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή Τροπολογία 11. Α, εδώ υπάρχει ένα λάθος. Οι 11 και οι 12 δεν είναι ασύμβατες. Μπορούν λοιπόν να συνδυαστούν. Η 12 δεν καταπίπτει εάν γίνει δεκτή η τροπολογία 11. Α, μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί. Όχι. Όχι. Την 11 θα ψηφίσουμε τώρα. Αρχικά υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Και η 12 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τελική ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή. Και τώρα θα ψηφίσουμε για τις γραμμές του προϋπολογισμού της τροπολογίας, οι οποίες είναι δύο. Η γραμμή είναι 20.0201 και είναι η 6777 υπέρ κατά αποχές δεκτή 67-78 τροπολογία υπέρ κατά αποχές το ίδιο αποτέλεσμα τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία και πέρας της ψηφοφορίας και δεκτεί με μία ψήφο κατά. Ε, συγχαρητήρια στον ε, Πίτερ Στάτσνη. Προχωρούμε τώρα στο σημείο 7 που είναι μία γνωμοδότηση με συντάκτη τον Τζο Χίγκινς από την ΚΟΕ για πτυχές αστικού, εμπορικού, γενιακού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης. Υπάρχουν εδώ κάποιες τροπολογίες και πρώτα θα ψηφίσουμε την πρώτη τροπολογία, τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. έλεγχος της ε, άρχιτη ψηφοφορία επί 1. Πέρας. Έλεγχος. Όχι, θα με τώρα. Άρχεται ψηφοφορία. Μπορώ να πω ότι τώρα είναι το πέρας της ψηφοφορίας, το είπα. Δεκτή λοιπόν. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Ψηφίζουμε την 9 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Α, ψηφίζομαι ηλεκτρονικά τη 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 10. Πέρας. Λειτουργήσε λοιπόν αυτή τη φορά το μηχανημά σας. Και τελική ψηφοφορία στο σχέδιο γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας και το αποτέλεσμα είναι θετικό. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στο Τζο Higgins. Περνάμε στο σημείο 8. για τις τροπολογίες για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ο Καντέρα Ρίφ είναι ο εισηγητής μας. Πρόκειται για γνωμοδότηση. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. Μία ψήφος μόνο κατά. Συγχαρητήρια κυρία Ρίφ. Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Πηγαίνουμε στο σημείο 9 τώρα για την υποχρεωτική εφαρμογή 69 κανονισμών της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με τις τεχνικές μονάδες που προορίζονται για τα οχήματα αυτά. Ο κύριος Καζά από τους φιλελευθέρους είναι ο εισηγητής μας. Στην ουσία θα γίνει μια πρώτη συζήτηση της σύστασης. Έχετε το λόγο κύριε Καζάκ. Ευχαριστώ πρόεδρε, συνάδελφοι. Όπως σωστά είπατε, πρόκειται για μια σύσταση την οποία σας καταφέτω που αφορά την υποχρεωτική εφαρμογή 61 κανονισμών της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την πιστοποίηση των αυτοκινήτων, των ρημουλκών και ε, των τεχνικών στοιχείων τα οποία υποχρεωτικά πηγαίνουν με αυτά και προορίζονται για αυτά. Αυτό θα έχει σαν στόχο την καλύτερη τεχνική συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Η ομάδα, η επιτροπή αυτή αποτελείται από 56 χώρες, τις οποίες προστίθενται ο Καναδάς, οι Ηνωμένε Πολιτείες, οι Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας και το Ισραήλ. Έχει σχέση με το περιβάλλον, το εμπόριο αλλά και ε, τις μεταφορές. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο προβλέπει την υποχρεωτική εφαρμογή των κανονισμών της Επιτροπής αυτής. Μέσα από την απόφαση του Συμβουλίου λοιπόν, οι 61 αυτοί κανονισμοί θα ενσωματωθούν στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αυτό θα μας επιτρέψει να μην υπάρχουν επικαλύψεις και σε τεχνολογικό επίπεδο και σε επίπεδο πιστοποίησης και σε επίπεδο διοικητικών διαδικασιών, κάτι το οποίο θα ωφελήσει τις βιομηχανίες αλλά και τον καταναλωτή. Και θα βελτιωθεί επίσης η πρόσβαση των προϊόντων αυτών σε τρίτες αγορές που έχουν προσυπογράψει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και της Οικονομικής της Επιτροπής του 1958 η βιομηχανία συμφωνεί με τις προτάσεις αυτές. Συνεπώς κύριε Πρόεδρε, σας προτείνω να δώσετε ένα συν στην πρόταση αυτή και μιας και εμείς επίσημα δεν έχει ζητηθεί η άποψή μας, σας προτείνω να ψηφίσουμε στην επόμενη συνάντηση, εφόσον βέβαια δεν έχουν υπάρξει εν μεταξύ προτάσεις αλλαγής των συγκεκριμένων κειμένων. Η, κανονικά η διαδικασία και η νομική βάση θα πρέπει να διευκρινιστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω της θέσης σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Επί τη βάση του άρθρου 81 του κανονισμού δεν είναι δυνατόν να κατατεθούν τροπολογίες στη συγκεκριμένη πρόταση. <laughs> Um, uh, Έχετε δίκιο παρατηρώντας ότι δεν έχουμε ακόμα έτοιμα επίσημο του Συμβουλίου, οπότε δεν ψηφίζουμε. Ήταν να ψηφίσουμε, αλλά δεν ψηφίζουμε. Θα περιμένουμε λοιπόν. Θα δώσω το λόγο στο Φλόραν Χέρλιτς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ευχαριστήσω τον κύριο Καζάκ για την παρέμβασή του και για την εξαιρετική δουλειά την οποία έκανε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δεν θα καθυστερήσω να θυμίσω μόνο ότι η πρωτοβουλία αυτή εγγράφεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, τον κανονισμό δηλαδή, για θέματα ασφαλείας 671, 661 μάλλον του 2009 που στην ουσία καθιστά υποχρεωτικές κάποιες ρυθμίσεις και κανονισμούς που προέρχονται από την Οικονομική Επιτροπή της Γενέβης εννοούμε των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι απλοποιούμε κάποιες παλαιότερες οδηγίες και διατηρούμε, ε, συμμορφούμε αν θέλετε, ε, στις ε, προτάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Δεν θα επαναλάβω τα υπό του κυρίου Καζάκλεχθέντα, αλλά θα ήθελα να πω ότι η πρωτοβουλία αυτή θα συζητηθεί στο Συμβούλιο ή μάλλον συζητήθηκε στο Συμβούλιο στις 27 Ιουλίου, έγινε μια πρώτη συζήτηση, δεν παρουσιάζονται ειδικέ δυσκολίες. Το θέμα της διευκρίνησης της νομικής βάσης δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Θα διευκρινιστεί στη συνάντηση του Συμβουλίου της 8 Σεπτεμβρίου και θα σας αποσταλεί το έγγραφο και θα μπορέσετε να ψηφίσετε εν γνώση των πραγμάτων αυτών. Ευχαριστώ. Κάποιο άλλο σχόλιο, κάποια άλλη παρατήρηση από τα μέλη. Όχι, συνεπώς. Σας ευχαριστώ κύριε Καζάκ. Περνάω στο 10, το οποίο είναι μια αντίστοιχη περίπτωση, υποχρεωτική εφαρμογή του κανονισμού αριθμός 100 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη για την έγκριση και των μηχανικίνητων οχημάτων σχετικά με την ηλεκτρική ασφάλεια. Ο Νικολό Ρινάλντι από τους Φιλελευθέρους έχει το λόγο. Να κάνουμε δηλαδή ό,τι κάναμε και στην περίπτωση του κυρίου Καζάκ. Ο κύριος Ρινάλντι έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι πιο εύκολη η περίπτωση η δική μου σε σχέση με το πακέτο του κυρίου Καζάκ που έπρεπε να εξετάσει 61 κανονισμούς. Εγώ έχω έναν κανονισμό και όλα είναι πολύ πιο εύκολα θα έλεγα προέρχεται από την ίδια πηγή ο κανονισμός αυτός, την Κοινωνική Επιτροπή που θέτει τεχνικά, ασφαλείας, τεχνικά επίπεδα ασφαλείας για τα υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όπως διευκρινίστηκε και από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντάσσεται στη νέα οδηγία πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόκειται για ένα μέσο απλούστευσης και διευκόλυνσης της παραγωγής ε, υβριδικών και ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ε, γιατί θα έπρεπε οι κατασκευαστές να προσφεύγουν σε διάφορες διαδικασίες πιστοποίησης, αλλά εδώ έχουμε όμως ε, ένα ενιαίο και μόνο μέσο δεν υπάρχει κανένα πολιτικό περιεχόμενο, εντάσσεται γενικότερα στις προσπάθειες που γίνονται για την μεγαλύτερη κυκλοφορία προϊόντων που μολύνουν λιγότερο, ε, αφορά την πράσινη οικονομία. Το πρόβλημα όπως και στην περίπτωση του κυρίου Καζάκ ε, προέρχεται από μας. Είναι το θέμα της νομικής βάσης, ισχύει ακριβώς το ίδιο και για μας. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα η νομική βάση. Δεν έχουμε ενημερωθεί ακόμα. Δεν έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς θα κάνουμε και γι' αυτό προτείνω και εγώ να εγκρίνουμε την πρόταση αυτή στην επόμενη συνεδρίασή μας, μιας και δεν θα υπάρχουν τροπολογίες και φυσικά προϋποτίθεται ότι δεν θα αλλάξει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Θέλει η Επιτροπή το λόγο. Κύριε Χέρλιτς, θέλετε κάτι να πείτε. Φυσικά. Βεβαίως. Να διευκρινίσω ότι σε αυτό τον κανονισμό δίνουμε λίγο μεγαλύτερη, αν θέλετε, σε εισαγωγικά ορατότητα. Θέλουμε εμείς να εμείνουμε στα ηλεκτροκίνητα οχήματα Πρόκειται για έναν κανονισμό ο οποίος είχε περιληφθεί και στην τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθαρή πράσινη οικονομία. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε τον μήνα Απρίλιο, τίποτα άλλο. Κάποιο άλλο μέλος θέλει να τονίσει κάτι. Ευχαριστώ κύριε Ρινάλντι. Δεν μας μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς ότι κολλησιεργούμε. Εμείς έχουμε προχωρήσει και περιμένουμε το Συμβούλιο. Τώρα περνάω στο σημείο 11. Μεταβατικές ρυθμίσεις για τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες ανάμεσα σε τρίτες χώρες και σε κράτη-μέλη. Πρόκειται για τον λεγόμενο grandfathering regulation, κανονισμό. Όπως γνωρίζετε η συνθήκη της Λισαβόνας δίνει νέες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απαιτείται ένας κανονισμός γύρω από την αντικατάσταση εκατοντάδων ε, τέτοιων επιμέρους ε, επενδυτικών συμφωνιών. Ο Σλίτερ είναι ο εισηγητής μας από τους Πρασίνους και του δίδω το λόγο. Πρόκειται για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, σημείο 11. Ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω όλους θερμά σε αυτήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, είναι μία από τις νέες μας εξουσίες. Οπότε βρισκόμαστε σε μία πρεμιέρα εδώ. Στις 7 Ιουλίου εκδόθηκε η ανακοίνωση και ήδη από εκεί φάνηκε ότι ίσως δημιουργηθούν προβλήματα σύγκρουση αρμοδιοτήτων. Αλλά τώρα έχουμε τη νέα συνθήκη που είναι σαφής ότι πρόκειται για κοινοτική αρμοδιότητα και θα πρέπει και τα τρία θεσμικά όργανα να συμφωνήσουν για το πώς θα το διαχειριστούν. Και μια και στο τρίγωνο αυτό της συναπόφασης βρίσκεται και το Κοινοβούλιο, έχουμε και εμείς το λόγο μας. Τώρα, αυτό για τις ε, τρέχουσες διμερείς συμφωνίες. Η Ευρωπαϊκή όμως ε, Ένωση πλέον αποκτά αρμοδιότητα και μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις νέες εξουσίες για να προχωρήσουμε ακόμη παραπέρα. Έχουμε πάνω από χίλιες διμέρειες συμφωνίες αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε μια νομική ασφάλεια και μια προβλέπεται συνύπαρξη, δηλαδή ισχύουν οι παλιές ε, συμφωνίες μέχρι ότου θεσπιστούν νέες. Καλή αυτή η συνύπαρξη, αλλά χρειαζόμαστε και μία ρήτρα λήξης σταδιακής εκπνοής, sunset clause. Μερικές από τις συμφωνίες αυτές είναι παμπάλες και θα πρέπει να εξυγχρονιστούν. Μερικές μάλιστα υιοθετούν και απεικιοκρατική προσέγγιση. Να φανταστείτε. Δηλαδή πάτε, φάτε και φύγετε ανεύθυνοι. Δεν είναι στοιχείο αυτό της νέας εμπορικής πολιτικής ένωσης. Δεν έχει καμία σχέση με την παλιά απεικιοκρατική πολιτική. Όλοι συμφωνούμε όμως ότι χρειάζεται πρώτα μια νομική ασφάλεια. Θα πρέπει να ξέρουμε που πατάμε, αλλά δεν μπορούμε να διονύσουμε την παλιά κατάσταση. Γιατί αν έχουμε χιλιάδες διαφορετικές εμπορικές συμφωνίες διμερείς με χώρες που είναι αντιφατικές μεταξύ τους, δεν μπορούμε να μιλούμε για μια ενιαία εμπορική πολιτική της Ένωσης. Οπότε αργά ή γρήγορα θα πρέπει να τεθεί ένα τέρμα σε αυτή την κατάσταση. Τώρα με τις επενδυτικές συμφωνίες έχουμε αυτό το grandfathering και τη μεταβατική περίοδο. Θα δούμε πόσο θα διαρκέσει και η δεύτερη έκθεση του Καντέρα Ρίφ μάλλον για την ε, συνολική επενδυτική πολιτική και το τρίτο τμήμα αφορά τις εντολές που θα πρέπει να λάβει η Επιτροπή από το Συμβούλιο και πώς θα αναμειχθεί το Συμβούλιο στις εντολές. Εμείς δεν θέλουμε να εκχωρήσουμε αρμοδιότητες για κανένα από τα τρία αυτά θέματα, γιατί η νέα επενδυτική πολιτική χρήζει νέας νομικής βάσης. Θέλουμε έναν εξυγχρονισμό, μια προσαρμογή προς τη νέα κατάσταση και δεν μπορούμε εμείς να αποποιηθούμε τον ευθυνό μας και να αφήσουμε όλες τις αρμοδιότητες στο Συμβούλιο και την Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα ή άλλες χώρες. Εμείς θέλουμε αρμοδιότητες και στους τρεις τομείς, όπως προβλέπει η συνθήκη. Η συνθήκη κατοχυρώνει τις αρμοδιότητες αυτές του Κοινοβουλίου, γι' αυτό και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Τώρα, ως προς το περιεχόμενο της πρότασης της Επιτροπής, όπως είπε και προηγουμένως, Έχουμε τις ε, παλιές διμερείς συμφωνίες. Μερικές ε, θα έρθουν σε αντίφαση με τη νέα εμπορική πολιτική της Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αποτρέψει μια τέτοια αντίφαση, να καραδοκεί ώστε να την εντοπίσει και θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι διατάξεις που θα ισχύσουν και οι κανόνες για τις νέες επενδυτικές εμπορικές συμφωνίες και να δούμε πώς θα εμπλακεί το, Κοινοβούλιο στη διαδικασία αυτή. Και μια και θα υπάρξει μια περίοδος συνύπαρξης του παλιού με το καινούριο, θα δούμε πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε την ε, ρήτρα του πλέον ευνοημένου κράτους, ευνοημένου κράτους αυτές τις συμφωνίες. Γιατί αν δίνουμε σε, σε μία χώρα κάποια δικαιώματα με βάση μια συμφωνία και δεν την έχει με βάση άλλη συμφωνία και θέλει να αξιοποιήσει τη ρήτρα του πλέον ευνοημένου κράτους, Μήπω μια τέτοια ρήτρα σε μια συμφωνία υπονομεύσει τη θέση μας σε άλλες συμφωνίες. Θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η κοινοτική στρατηγική απέναντι σε αυτό το θέμα. Και αυτό το ζήτημα θα πρέπει να το διαθετήσουμε και για τη μεταβατική περίοδο, αλλά και για τη διαμόρφωση τη νέα μα εμπορική στρατηγική. Επίση χρειαζόμαστε κάποιε ελάχιστε προδιαγραφέ για τι επενδυτικέ συμφωνίε. Για παράδειγμα, διαφάνεια στο διακανονισμό των διαφορών. Και αυτό το ζήτημα είναι κάπω θολό αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αδιαφανεί και απόρριτε διαδικασίε ε, για κάποια πάνελ που λαμβάνουν αποφάσεις πολύ σημαντικές θα πρέπει αυτή η αδιαφάνεια να παταχθεί. Χρειαζόμαστε διαφάνεια στις συμφωνίες αυτές και να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των επενδυτών. Επίσης, μια συνολική πολιτική προϋποθέτει μια συνέπεια και μια συνάφεια. Δεν μπορούμε να απαιτούμε περιβαλλοντικές και κοινωνικές προδιαγραφές της νέας μας συμφωνίες και να συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε συμφωνίες με άλλες χώρες που παραβιάζουν τέτοιου είδους προδιαγραφές. Επαναλαμβάνω, μερικές από τις εμπορικές μας συμφωνίες είναι παμπάλες και είναι τελείως άσχετες με τους ε, νέους στόχους της ε, κοινοτικής εμπορικής πολιτικής. Και ίσως και χώρες όπως η Γερμανία, οι κάτω χώρες, η Μεγάλη Βρετανία έχουν ήδη πολλές διμερείς συμφωνίες με τις χώρες αυτές, με παλιές χώρες, αλλά νέες χώρες δεν έχουν τέτοιες συμφωνίες. Οπότε και εδώ θα πρέπει να δούμε πώς και οι νέες χώρες θα μπορούσαν να συνάψουν τέτοιες συμφωνίες. Να αποφευχθούν ανισορροπίες. Επίσης, εξασφάλιση ηθικών ίσου ανταγωνισμού για όλες τις ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί η μεταβατική περίοδος μπορεί να διαρκέσει αρκετά. Δεν θέλουμε ανισότητα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς ίσως μεταβατικής περίοδου. Και υπάρχουν κάποιες προβλέψεις για την αναθεώρηση. Λέμε το αργότερο πέντε χρόνια μετά τη θέση ισχύ του κανονισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει την ανάγκη για την συνέχιση ε, της εφαρμογής και την επαναδιαπραγμάτευση από τα κράτη-μέλη ή τη σύναψη νέων συμφωνιών. Δυστυχώς δεν υπάρχει πρόταση για μια ρήτρα εκπνοής, sunset clause. Θα πρέπει να υπάρξει μια ημερομηνία σταδιακής έστω αλλά εκπνοής, γιατί αν δεν έχουμε μια τέτοια καταληκτική προθεσμία, ποτέ δεν θα τεθεί ένα τέρμα σε αυτό το χαοτικό δεσμευτικό καθεστώς των χιλιάδων διμερών συμφωνιών. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για να θεσπίσουμε μια τέτοια ρήτρα εκπνοής. Έχουμε τη νέα συνθήκη της Λισαβόνα. θα πρέπει να τη σεβαστούμε και η πληθώρα αυτών των παλιών εμπορικών συμφωνιών δεν συνάδει με τη συνθήκη. Και μάλιστα η ύπαρξή του υπονομεύει και τη μελλοντική μα εμπορική πολιτική. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα τη συζήτηση που θα γίνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίζει και κάποιες νομικές πτυχές στις συμφωνίες. Άρθρο 9α, β και γ. Για παράδειγμα, σε ό,τι φορά το κοινοτικό δίκαιο, φυσικά όλες οι συμφωνίες θα πρέπει να τηρούν το κοινοτικό δίκαιο και υπάρχει το θέμα της επικάλυψης με διάφορε διάφορες νομοθετικές διατάξεις. Είναι πιο τυπικά νομικά ζητήματα στο σημείο Γ, κάτι πολύ ενδιαφέρον, 9 Γ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει την έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων, εκτός και αν θεωρήσει ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων αντιβαίνουν σε κάποιες νομοθετικές διατάξεις ή, λέει το ΓΑΜΑ, ε, δημιουργούν κόλλημα στην ανάπτυξη ή την εφαρμογή της ε, επενδυτικής κοινωνικής πολιτικής, ιδιαίτερα της κοινή εμπορικής πολιτικής. Εδώ δεν μου αρέσει αυτό που λέμε όλες οι κοινωνικέ πολιτικές που αφορούν τις επενδύσεις, γιατί αυτή είναι η ιδέα της σύγχρονης εμπορικής πολιτικής. Είναι ότι συμπεριλαμβάνει τις επενδύσεις ως ε, μέσο για την υλοποίηση άλλων κοινωνικών και περιβαλλοντικών σκοπών. Αυτή είναι η σύγχρονη εμπορική πολιτική. Αλλά λέμε που σχετίζονται μόνο με τις επενδύσεις, όπως λέει το γάμα στο 9, θα μπορούσαμε να θετήσουμε μια διασταλτική ερμηνεία, αλλά θα μπορούσαμε να θετήσουμε και συσταλτική ερμηνεία, οπότε θα πρέπει να το προσδιορίσουμε. Εγώ προτιμώ διασταλτική ερμηνεία, δηλαδή για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Αυτός είναι και ο σκοπός της σύναψης των συμφωνιών. Οπότε και αυτό θα ήθελα να το εξετάσουμε. Αυτά προς το παρόν και περιμένω τις ε, απόψεις των συναδέλφων Υπολογίζω στη συνεργασία σας και μην διστάστε. Αν έχετε προτάσεις, παρακαλώ να τις υποβάλλετε το συντομότερο δυνατό, όσο, το, όσο νωρίτερα, τόσο το καλύτερο, για να συμπεριληφθούν από την αρχή στο σχέδιό μου. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ανάλυση του κανονισμού και τα προβλήματα, τα θέματα που θέτει και που πρέπει να θέτει. Πριν δώσω στην Κομισιόν και το Συμβούλιο το λόγο, ας ακούσουμε τις άλλες πολιτικές ομάδες. Ο κύριος ε, Καλύφ. Ευχαριστώ. Δεν έχω να προσθέσω και πολλά. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σλέτερ γιατί έκανε μια γενική επισκόπηση του προβληματισμού για αυτές τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες. Τον Ιούλιο είχαμε μια συζήτηση για κλεισμένο το θηρό με τον κύριο Σάλιβαν και το ανέφερε αυτό και ο κύριος Σλέτερ. Το θέμα των επενδυτικών συμφωνιών θα αποτελέσει σημαντικό τμήμα του έργου της Επιτροπής μας τους επόμενους μήνες. Είναι πολύ ευαίσθητο αυτό το θέμα και μάλιστα η συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει σημαντικές αρμοδιότητες για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να τις αξιοποιήσουμε στο έπακρο. ιδιαίτερα για το θέμα των επενδύσεων. Μας είπαν ότι οι μεταβατικές διατάξεις θα υιοθετηθούν με τη διαδικασία συναπόφασης. Οπότε το Κοινοβούλιο θα συμμετέχει εκεί. Αλλά μας είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται και νέες επενδυτικές συμφωνίες με την Ινδία, τον Καναδά, τη Σιγκαπούρη, με το Μερκοσούρ, με πολύ σοβαρές συνέπειες. Εκεί έχουμε την ε, αίσθηση ότι μας παραγκώνησε κάπως, παραμέρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε, τι γίνεται. Οι διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες ε, δεν θα πρέπει να ξεκινήσουν αν δεν υιοθετηθεί η έκθεση η πρωτοβουλία του Συμβουλίου με τη θέση του Συμβουλίου. Επίση, η Συμφωνία Πλαίσιο Κοινοβουλίου Επιτροπή υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε διαπραγματευτική εντολή θα πρέπει να αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα σε μια προθεσμία που θα επιτρέψει την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των βουλευτών. Ελπίζω να τηρηθεί αυτή η συμφωνία και να λάβουμε το συντομότερο δυνατό το σχέδιο διαπραγματευτικής εντολή για τι διαπραγματεύσεις με τις τρίτες χώρες ε, για τα επενδυτικά θέματα. Αυτά, ευχαριστώ. Yeah. Ε, Ευχαριστώ κύριο Κάσπαρη. Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα του κυρίου Αρίφ για τις συμφωνίες που θα διαπραγματευτούμε με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Τονίζω όμως την έκθεση του συναδέλφου Σλούτερ που συζητούμε σήμερα. Δεν είμαι ικανοποιημένο από το σχέδιο που υπέβαλε η Κομισιόν. Είμαι πεισμένο ότι δημιουργείται μεγάλη νομική αβεβαιότητα μεταξύ επενδυτών στην βιομηχανία. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις σχετικά με το τι θα γίνει αν προσβληθούν οι συμφωνίες και αν ε, γίνει προσφυγή σε δικαστήρια ή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με βάση τις συμφωνίες αυτές. Αυτό δεν είναι καλό ούτε για τις θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, ούτε για τους αναπτυξιακούς στόχους που ανέφερε ο κ. Φλούτερ. Και αν σκεφτούμε και τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στο εξωτερικό που ε, είναι μακράς πνοής, ε, ως επιτοπλίστων δεν θέλουμε μία ε, εφάπαξ ε, εξέταση των συμφωνιών που θα διακινδυνεύσει τις επενδύσεις μας. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσουμε πολύ συγκεκριμένα τις υφιστάμενες συμφωνίες με το Sunset Clause. Κάποια στιγμή όλες οι συμφωνίες εκπνέουν. Ε, οπότε εδώ πιστεύω ε, ότι εδώ χρειάζεται νομική βεβαιότητα για τις επιχειρήσεις, για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών απέναντι στους διεθνείς εταίρους μας. Αυτό πρέπει να είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας. Γι' αυτό το θέμα sunset clause, ρήτρα εκπνοής, θα πρέπει να το εξετάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά. Δεν ε, το αντιμετωπίζει σωστά η Κομισιόν. Και κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι αν η Κομισιόν θέλει να διαπραγματευτεί στο μέλλον νέα συμφωνία, προτείνει σε εκείνη την περίπτωση να μην δοθεί από το Συμβούλιο έγκαιρα εντολή για την ε, δήλωση ε, ότι είναι άκυρες οι συμφωνίες. Μπορεί δηλαδή εδώ να ασκηθεί κάποιος εκβιασμός, μπορεί δηλαδή και η Κομισιό να μπορεί να εκβιάζει το Κοινοβούλιο ούτως ώστε να ε, δίδει εντολές και μπορεί με κάποια, σε, κάποια ε, χώρα να μην υπάρξει τέτοια συμφωνία για κοινωνικούς λόγους, για λόγους ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Να μην θέλουμε και μπορεί η Κομισιόν να ασκήσει εκβιαστικά πιέσεις ε, ε, και θα πει ότι ε, αν δεν δώσει εντολή το Συμβούλιο μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε διότι δεν θα υπάρχει εντολή. Ε, είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ε, δούμε εντατικά, ε, μέσα από εντατικές συζητήσεις το θέμα και μέσα από ένα χρονοδιάγραμμα να καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική λύση για την ψηφοφορία, ούτως ώστε να έχουμε χρόνο μεταξύ ψηφοφοριών, τροπολογιών, τελικών κειμένων, ώστε να έχουμε χρόνο να επεξεργαστούμε συμβιβαστικές προτάσεις με την ησυχία μας και παρακολουθώντας όλα τα θέματα και τις πτυχές. Ευχαριστώ πολύ. Από την ομάδα των φιλελευθέρων, η κυρία Τεσάρνης. Ευχαριστώ. Από τους φιλελευθέρους λοιπόν και δημοκράτες. Θα συμφωνήσω με τους τρεις προλαλήσαντες. Το θέμα όμως τίθεται και με διαφορετικό τρόπο και το λέω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλό είναι να θέτει κανείς το θέμα των μεταβατικών ρυθμίσεων και κατανοώ το θέμα της νομικής αβεβαιότητας που δεν θα πρέπει να μας χαρακτηρίσει. Αλλά το να θέσει το θέμα των μεταβατικών ρυθμίσεων χωρίς να θέσουμε τον βασικό στόχο, το ποιο είναι ο στόχος μας, ποια είναι η πολιτική μας και ποια είναι ακριβώς η πολιτική την οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε προκαταλαμβάνουμε τις καταστάσεις χωρίς να γνωρίζουμε το τι θα ακολουθήσει. Λοιπόν, δεν πάει έτσι το πράγμα, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εκθέτει και αν η συνθήκη της Λισαβόνας έχει κάποιο νόημα και αν εμείς έχουμε κάποιες υποχρεώσεις σύμφωνα με αυτήν, το θέμα είναι να θέτουμε τα πράγματα ε, επί της ουσίας η ουσία λοιπόν δεν είναι οι μεταβατικέ ρυθμίσει, αν και η έκθεση είναι σημαντική, αλλά το θέμα είναι τι είδου επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να κάνει, τι σχέσει θέλει να έχει με τι τρίτε χώρε, τι σχέσει στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντο των κοινωνικών δικαιωμάτων. Εγώ θα ήθελα δηλαδή να καθορίσουμε τον στόχο και τη στρατηγική πριν ασχοληθούμε με θέματα πρακτικά χρονοδιαγράμματος. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο η παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ. I think I should preface my... Πια σήμερα. Λοιπόν, ε, σας εκτιμώ τους περισσότερους από σας εγώ ήρθα εδώ όμως για να προστατεύσω τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι τα συμφέροντα ενός ευρωπαϊκού υπερκράτους. Και όταν βλέπω τις προτάσεις αυτές από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου, τότε πραγματικά ανησυχώ ιδιαίτερα. Λέγει εδώ η πρόταση ότι η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει την αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις άμεσες επενδύσεις τις εξωτερικές. Αποκλειστικές αρμοδιότητες, τα επαναλαμβάνω αυτά γιατί τα επαναλαμβάνει το κείμενο. Ο κύριος Σλάιτα, ο οποίος ε, είναι ιδιαίτερα κομψός στα επιχειρήματά του, πάρα πολύ σωστά και ακριβέστατα είπε ότι υπάρχουν χιλιάδες διμερείς συμφωνίες επενδυτικές ανάμεσα ε, στα εθνικά επίπεδα. Κάποιες χώρες έχουν ε, εκατοντάδες, κάποιες έχουν επίσης πολύ λίγες τέτοιες συμφωνίες. Και είπε επίσης ο κύριος Σλούτερ και εδώ διαφωνώ ότι δεν μπορεί να υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα οι διαφορετικές χώρες, τα διαφορετικά μέλη είναι ακριβώς διαφορετικά. Δεν είναι το ίδιο. Δεν πιστεύω σε αυτή την ψευδέστηση στο ότι όλοι είμαστε ίδιοι ενώ είμαστε όλοι διαφορετικοί. Μία από τις χώρες λοιπόν που έχει πάρα πολλές διμερείς συμφωνίες είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Το 40% όλων των διμερών επενδυτικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση περνά από το Ηνωμένο Βασίλειο, έρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και σχετικά με τις έκροες, σε αυτή την περίπτωση το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία από τις μεγαλύτερες επενδύτριες χώρες. Παράδειγμα, όπως και οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας και επενδυτής στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στις Ηνωμένε Πολιτείε. Με τα στοιχεία αυτά λοιπόν και όταν φτάνει κανείς στο κεφάλαιο 3 και βλέπει τι λένε όλες αυτές οι ρήτρες, το άρθρο 8 λέει σαν παράδειγμα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει όταν ένα κράτος θέλει να τροποποιήσει μια συμφωνία ή να συνάψει μια νέα τέτοια διμερή συμφωνία. Το άρθρο 9 καθορίζει τις λεπτομέρειες επί τη βάση των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα επιτρέψει την έναρξη των διαπραγματεύσεων από τα κράτη-μέλη με τρίτες χώρες για τη σύναψη μιας νέας συμφωνίας. Το άρθρο 10 λέγει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν συστηματικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή μπορεί επιπλέον να ζητήσει να πάρει μέρος στις διαπραγματεύσεις αυτές σαν παρατηρήτρια. Στο άρθρο 11 για την εφαρμογή της συμφωνίας η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα αξιολογήσει ότι δεν υπονομεύει αντίστοιχες διαπραγματεύσεις εμπορικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να βρίσκονται σε αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Λοιπόν, όλες αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές οι οποίες είναι ιδιαίτερα βλαβερές από την για την χώρα μου ο Ντέβιτ Μάρτιν ε, τον βλέπω να χαμηλοβλεπεί ουσιαστικά. Πού ήταν ο Ντέβιτ Μάρτιν όταν δέχτηκε τη συνθήκη αυτή χωρίς ε, καθόλου επιφυλάξεις. Εγώ τους περισσότερους συναδέλφους τους αγαπώ και τους σέβομαι. Αλλά παρόλα αυτά η προοπτική αυτή η οποία μας ανοίγεται είναι μια τρομακτική προοπτική για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ιδιαίτερα για τον επιχειρηματικό κόσμο την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου. Νομίζω ότι στην ουσία στο μέλλον ένας γαλλογερμανός πράσινος θα έχει δικαίωμα κυρίας σε επενδυτικές προσπάθειες που θα δημιουργούν θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο υποφέρει από συστηματικές παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομία μας έχει επιβαρυνθεί από απαράδεκτες νομοθετικές ρυθμίσεις και νομίζω ότι κάποιες από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός ε, της δικής μου το νιώθουν αυτό. Οι προτάσεις αυτές λοιπόν δεν είναι παραπρόδρομος, κάτι το οποίο θα είναι ιδιαίτερα βλαβερό και ε, γι' αυτό ακόμα και όταν ε, οι βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου αποστρέφουν το βλέμμα τους όταν τα λέω αυτά, θα έρθει η ώρα που θα μετρηθούν όλοι. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Πετριτσιόνε, από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Δεν θα μιλήσω γενικόλογα για τη σημασία των επενδύσεων. Τρία πράγματα θα κάνω. Θα θυμίσω πώς βλέπει η Κομισιόν τη νέα πολιτική μέσα στο πλαίσιο της κοινή εμπορικής πολιτικής. Το σκεπτικό γιατί υποβάλαμε το συγκεκριμένο έγγραφο και σύντομα θα υπενθυμίσω τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδίου κανονισμού που ελπίζω ότι θα αρχίσουν να απαντούν σε κάποιες ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής, αν και πρέπει να πω ότι πολλά από τα θέματα αυτά είναι περίπλοκα και δεν ισχυρίζομαι ότι σε αυτό το στάδιο μπορώ να απαντήσω σε όλα. Κύριε Πρόεδρε, γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι πολιτικές μας ε, ε, εγγυώνται ότι ότι θα έχουν ε, ε, ίσους κανόνες ε, παιχνιδιού οι επενδυτές και για τη λειτουργία τους στην αγορά. Ο όλος σκοπός των επενδύσεων στα πλαίσια της κοινή εμπορικής πολιτικής είναι για να υπάρχει παρόμοια μεταχείριση των Ευρωπαίων επενδυτών στο εξωτερικό ε, σε σχέση με τους ξένους στην Ευρώπη. Οι, διαπραγμα... συμφωνίες ε, επενδύσεων δεν ε, παρακάμπτουν την... το δίκαιο είτε στην Ευρώπη είτε στο... το... το δίκαιο των εταίρων. Αυτό είναι η προϋπόθεση για τις νέες διατάξεις κατά τη γνώμη της Κομισιόν στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι πολύ σημαντικό και το γνωρίζει απόλυτα η Κομισιόν να σημειώσουμε ότι έτσι η επενδυτική πολιτική ε, μπαίνει μέσα σε συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο και το βασικό χαρακτηριστικό του νέου θεσμικού πλαισίου είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Η Κομισιόν έχει δεσμευτεί απόλυτα να παίξει το ρόλο της ε, ως προς αυτό. Όπως αναφέρθηκε, όταν αναπτύσσουμε νέα πολιτική δεν αγνοούμε το γεγονός ότι έχουμε 1.200 διμερείς συμφωνίες επενδύσεων από τα κράτη, που έχουν συναυθεί από τα κράτη-μέλη. Και επειδή δεν υπάρχουν κοινοτικές ή ενωσιακές συμφωνίες, αυτές είναι οι συμφωνίες που προστατεύουν τους επενδυτές στο εξωτερικό και διασφαλίζουν στους ξένους επενδυτές ότι η πολιτική μας απέναντί τους δεν θα αλλάξει ε, άρδιν διαχρονικά. Αυτή η συμφωνία παραμένει ενισχύει στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αν δεν αλλάξει τίποτα παραμένουν ενισχύει και υπάρχει νομική βεβαιότητα έτσι στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Το πρόβλημα είναι ότι η σύγκρουση με τις αποκλειστικές δραστηριότητες, ε, ε, ε, θέτει ένα αμφιβόλο το δικαίωμα των κρατών μελών να ε, προσβάλλουν τις ε, συμφωνίες και αυτό θέλουμε να αλλάξουμε. Θα πρέπει να υπάρχει χρόνος να περάσουμε τη θεσμική διαδικασία έγκρισης αυτού του κανονισμού που θα πάρει όσο χρόνο χρειαστεί στα πλαίσια της νομοθετικής διαδικασίας. Είναι σημαντικό να ε, έχουν, να πάρει ένα μήνυμα οι επενδυτές, ξένοι επενδυτές, ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης λειτουργούν για να διορθωθούν αυτά τα θέματα. Ταυτόχρονα, ήδη σήμερα έγινε η παρατήρηση για τη νομική βεβαιότητα που θα διασφαλιστεί ε, διατηρώντας ε, προς το παρόν το κεκτημένο που υφίσταται και ότι αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν προδικάζει τη μελλοντική πολιτική ο, της Ένωσης ο κανονισμός. Θα πρέπει να τηρηθεί το γράμμα και το πνεύμα της συνθήκης. Υπάρχουν πολλές ε, διατάξεις στον κανονισμό που σκοπό έχουν να επιτύχουν ακριβώς αυτό το στόχο. Η συζήτηση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα δείξει αν τα καταφέραμε, αλλά ο στόχος αυτός ήταν. Ταυτόχρονα, και γι' αυτό η Κομισιόν έκανε την ε, ανακοίνωση για τη μελλοντική επενδυτική πολιτική. Αυτή η ανακοίνωση πρώτο βήμα είναι, δεν απαντά σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά τουλάχιστον σηματοδοτεί ότι θα εξελιχθεί η πολιτική και κάποιες αδρές γραμμές ε, τίθενται. Αναφέρεται ότι η εξέλιξη θα είναι σαφή, σταδιακή, προβλέψιμη, θα στηρίζεται σε μια διαφανή αντιπαράθεση μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των εμπλεκομένων και θέτει κάποιες βασικές αρχές για τις πολιτικές επιλογές που θα αντιμετωπίσουμε ενδεχομένω πολύ πρόθεσμα. Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία αυτού του κανονισμού, κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, ο κανονισμός θέλει να ε, τονίσει την νομιμότητα της ύπαρξης αυτών των συμφωνιών. Ε, δεν αποτελεί πατρογονική ρήτρα σε καμία. Οποιαδήποτε παραβίαση της συνθήκης ε, δεν μπορεί να καλυφθεί από το συγκεκριμένο κανονισμό, ο οποίος λέει ότι η έγκριση δεν παραβλάπτει την υποχρέωση των κρατών μελών στα πλαίσια της συνθήκης. Παραμένουν απόλυτα υπεύθυνα για την απάλληψη οποιασδήποτε συμβατότητας και η Κομισιόν διατηρεί τη νομική αρμοδιότητα να αναλάβει νομική δράση, αν κρίνει σκόπιμο. Δεν προτιθέμεθα με τον κανονισμό αυτόν να αλλάξουμε τα νομικά δεδομένα πέρα από την κατάργηση σε προσωρινή βάση της ασυμβατότητας που δημιουργείται από το θέμα της ε, αρμοδιότητας. Δεύτερον, η εξουσιοδότηση των κρατών μελών να συνεχίζουν να διαπραγματεύονται διμερείς συμφωνίες. Αυτό είναι εξαιρετική συμφωνία, περιορισμένη χρονικά και ως προς το πεδίο εφαρμογής περιορισμένη. Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι αυτό το μηχανισμό. Πρώτον, η δημιουργία ενωσιακής πολιτικής θα είναι, υποχρεωτικά θα είναι σταδιακή. Ακόμα και αν είχαμε τους απαραίτητους πόρους και την απαραίτητη γνώση, θα ήταν αντικειμενικά δύνατον η Ένωση να αντικαταστήσει 1.200 συμφωνίες ε, σε οποιοδήποτε εύλογο χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν η θέσπιση ενουσιακής πολιτικής θα είναι σταδιακή, αυτό είναι αναπόφευκτο και ο μεταβατικός ε, μηχανισμός ε, σκοπό έχει να αμβλύνει τα αρνητικά αποτελέσματα αυτής της σταδιακής εξέλιξης. Η εξουσιοδότηση για επαναδιαπραγμάτευση των κρατών μελών και αυτή δικαιολογείται. πολλέ από αυτέ οι συμφωνίε, είναι πολλέ παλιέ είναι πολύ παλιές, αλλά έχουν ε, ρήτρες ανανέωσης και ανανεώνονται, θέλουμε να ανανεώνονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και έτσι περνώ στο δεύτερο λόγο εξουσιοδότησης. Πολλές από αυτές τις συμφωνίες έχουν πολλές ασυμβατότητες με τη συνθήκη και τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να το διορθώσουν αυτό. Η εξουσιοδότηση της αναδιαπραγμάτευσης τους το επιτρέπει αυτό. Είναι ένα μέσο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη ούτως ώστε να λύσουν το θέμα της σημαντικής ασυμβατότητας που πολλές φορές έχει εντοπιστεί και από το δικαστήριο. Το τρίτο στοιχείο που τονίζω και αυτό είναι το τελευταίο σημείο που θέλω να αναφέρω σε σχέση με τον κανονισμό η ρήτρα ανάκλησης και αναθεώρησης η επανεξέταση. Θέλαμε να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και ακριβείς σχετικά με τους λόγους ανάκλησης της έκδοσης ε, ή της απόρριψής της. Προφανώς ε, οι λεπτομέρειες θα συζητηθούν και εδώ και στο Συμβούλιο. Θέλαμε να είμαστε όσο γίνεται ακριβέστεροι. Έχω καταγράψει κάποιες επικρίσεις σας. Παραμένει όμως γεγονός ότι αν κάποια συμβατότητα προκύψει σε σχέση με τη συνθήκη, τότε η Κομισιόν οπωσδήποτε χρειάζεται να έχει την εξουσία να σταματήσει την ε, επαναδιαπραγμάτευση ε, η ανανέωση αυτής της ε, συμφωνίας. Δεν θα προσφύγομαι στο δικαστήριο, γιατί παίρνει χρόνο, αν, αν δηλαδή έχουμε ταχύτερο μέσον στα χέρια μας, προβλέπεται και διαβούλευση που μας, θα μας επιτρέπει να λύνουμε τα προβλήματα σε διαβουλεύσεις με το ενδιαφερόμενο κάθε φορά κράτος μέλος. Παραμένει όμως γεγονός ότι τώρα υπάρχει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε ένα προσωρινό μηχανισμό εξαιρετικό. Εάν αποδειχθεί ότι ο μηχανισμός εξουσιοδότησης συγκρούεται με την ενωσιακή πολιτική ανάπτυξη, η Κομισιόν θα πρέπει να έχει την εξουσία να το πει αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν αρκετές νομικές εγγύησεις για να αποφευθούν οι καταχρήσεις. Ε, τέλος, τελευταία παρατήρηση αφορά κάποια από τα θέματα που έθεσαν τα μέλη της Επιτροπής σας. Προσπαθούμε να υποβάλλουμε ένα πακέτο εγγράφων και μέσων που θα δίνει όσο γίνεται πληρέστερη εικόνα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εικόνα που μπορεί να έχει η επενδυτική πολιτική. Είναι πλήρης εικόνα? Όχι. Δεν έχουμε όλα τα στοιχεία άλλωστε για να, σα να, δώσουμε, ε, να σας δώσουμε πλήρη εικόνα. Ούτε εμείς δεν έχουμε. Κάνουμε όμως ό,τι είναι δυνατόν για την πληρότητα Έχουμε διαπραγματευτικές εντολές για την απελευθέρωση των επενδύσεων σε όλες τις διαπραγματεύσεις σχεδόν που ε, ενέχεται και συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε όμως εντολή για την προστασία των επενδύσεων. Καμιά φορά οι εμπορικοί εταίροι μας ε, έκαναν προϋπόθεση την προστασία των επενδύσεων για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, οι εμπορικές. Και είναι αδιανόητο να μην διαπραγματεύεται η Ένωση ένα σημαντικό θέμα με τους εταίρους, όπως θα ήταν αδιανόητο να μας έλεγαν και εκείνοι κάτι που ενδιαφέρει πολύ εμάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν ολοκληρωθεί. Η Κομισιόν θέλει να ζητήσει ε, μια οδηγία συμπληρωματική για τη διαπραγμάτευση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα για να μπορέσει να το χειριστεί. Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα ολοκληρωθούν αύριο. Θα εκπλαγώ αν οι διαπραγματεύσεις ε, ε, όχι, δεν θα, θα τελειώσουν αύριο, θα ε, μου κάνει έκπληξη αν ε, ολοκληρωθούν πριν ολοκληρώσει τις διαδικασίες του Κοινοβούλιο. Η ό,τι αφορά τις νέες διαπραγματεύσεις και τώρα διερευνούμε αν θα είχε νόημα να γίνει μια επένδυση με την Κίνα, αυτό σημαίνει ότι θα γίνει αξιολόγηση το, των επιπτώσεων, δημόσια διαβούλευση, η εντολή θα παρουσιαστεί στο Κοινοβούλιο από την Κομισιόν όλες οι εντολές παρουσιάζονται στο Κοινοβούλιο, έτσι προβλέπει η Συμφωνία Πλαίσιο άλλωστε, και μετά θα δούμε αν θα λάβουμε καταρχήν την εντολή. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία είναι αρκετά χρονοβόρα επίσης και δεν προβλέπουμε ότι θα προδικάσει κατιονδήποτε τρόπο τις συζητήσεις που θα γίνουν στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις αδρές γραμμές της πολιτικής. Και τέλος, Πιστεύουμε ότι θα βοηθούσε επίσης και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να έχουν τουλάχιστον μερικά συγκεκριμένα ε, παραδείγματα σχετικά με το πώς θα μπορούσε να είναι η προστασία των επενδύσεων καθώς θα συζητούν το κανονισμό και την ανακοίνωση. Δεν μπορέσαμε να παρουσιάσουμε στην ανακοίνωση το τρόπο αυτό, το μέσο αυτό, ε, με αφηρημένο τρόπο, αλλά θα μιλήσουμε για συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου θα πρέπει να συζητήσουμε με τους εταίρους μας και πιστεύουμε ότι αυτό θα τροφοδοτήσει τη συζήτηση αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Και τώρα από το Συμβούλιο. Ο κύριος Κάσπαρ. Συμπληρωματική ερώτηση προς την Κομισιόν, αφού εκπρόσωπος της Κομισιόν ασχολήθηκε ε, εντελεχώς με το θέμα. Η συμπληρωματική ερώτηση είναι η Ε, Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν μίλησε για τις υφιστάμενες συμφωνίες και σε ποιο βαθμό συγκρούονται με τη, συμφωνία, με τη συνθήκη. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται αρμόδια για τη διαπραγμάτευση και όχι πια τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Δεν είμαι νομικός, αλλά και ο πρόεδρος γνωρίζει ότι η Κομισιόν πάντα ήταν ο θεματοφύλακα των ευρωπαϊκών συνθήκων. Και αυτό που είναι μυστηριώδες για μένα είναι γιατί η Κομισιόν προφανώς τι τελευταίες δεκαετίες το θέμα αυτό των χιλίων και πάνω ε, συμφωνιών που ε, μπορεί να παρουσίαζαν πρόβλημα, όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν δεν ασχολήθηκε με αυτές. Αν δηλαδή ήταν είτε είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα είτε δεν είναι το θέμα αυτό, η Κομισιόν είναι αρμόδια να φροντίζει ούτως ώστε να μην συνάπτονται συμφωνίες που συγκρούνται με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δηλαδή, κοιμόταν τις τελευταίες δεκαετίες η Κομισιόν. Εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι. Υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα που πριν από την 1η Δεκεμβρίου δεν υπήρχαν. Γιατί δηλαδή τώρα ξαφνικά θα πρέπει να επαναξεταστούν όλες οι συμφωνίες προστασίας των επενδύσεων ενώ ε, αυτό δεν γινόταν παλιά ενώ παρόλα αυτά θα έπρεπε οι συνθήκες να τηρούνται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει. Ευχαριστώ. Υπάρχει ρήτρα διαφάνειας και σκοπός της είναι να αποφύγει η επανάληψη της κατάστασης των τελευταίων 20 ετών, όπου είχαμε πολύ αμυδρή ιδέα για το ότι περίχανε συμφωνίες, γιατί τα κράτη-μέλη δεν είχαν υποχρέωση να κοινοποιήσουν τις συμφωνίες αυτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να τις δείξουν σε οποιονδήποτε. Παρ' όλα αυτά προσφύγαμε στο δικαστήριο κατά πολλών χωρών για συμβατότητα με τη συνθήκη. Και μάλιστα μερικές φορές οι διαπραγματεύσεις βέβαια συνάπτονταν καλόπιστα ή τουλάχιστον οι διαπραγματεύσεις γίνονταν καλόπιστα. Δεν λέω ότι τα κρατημέλη ε, εσκεμμένα διαπραγματεύοντα συμφωνίε που γνώριζαν τα ασύμβατες με τη συνθήκη, αλλά ανέκυψε το θέμα τη ασυμβατότητα στην πορεία. Και όταν το έμαθε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέλαβε δράση, είτε πείθοντα τα κράτη-μέρη να επαναδιαπραγματευτούν τι συμφωνίε. Και μάλιστα στη διεύρυνση του 2004 έγινε εγχείρημα παρόμοια μεγάλης εμβέλειας και πολλές προσπάθειες αναδιαπραγμάτευσης ακριβώς για να αποφευθούν οι συμβατότητες με τη συνθήκη στα πλαίσια της, διαπρα... του 2004 και εκεί που υπήρχε διαφωνία μεταξύ χώρας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασυμβατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέφυγε στο δικαστήριο κατά της ε, λόγω χώρας. Ήταν πολλές οι συμφωνίες, καμιά τετρακοσαριά Τι ε, εξετάσαμε ενδελεχώς και φυσικά για να αρθούν όλες οι αβεβαιότητες ε, θα χρειαστεί καιρό. Οπότε ο νέος μηχανισμός μας εφοδιάζει με νέα εργαλεία για την διόρθωση της ασυμβατότητας σε περίπτωση που εντοπιστεί. Υπάρχει και ένας μηχανισμός διαβούλευσης που προβλέπεται, ώστε όταν στην αναδιαπραγμάτευση μια τέτοια συμφωνία κατά τη μεταβατική περίοδο το κράτος μέλος μπορεί σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει διόρθωση της ασυμβατότητας χωρίς να αφισβητείται η ισχύ της συνθήκης κάτι που θα ήταν εις βάρος της σταθερότητας που όλοι επιθυμούμε. Εγώ δεν λέω ότι είναι τελείως ε, άψογος αυτός ο μηχανισμός, ότι είναι αψεγάδιαστος και ότι θα λειτουργήσει απρόσκοπτα και χωρίς κανένα πρόβλημα, αλλά φροντίζουμε και με άλλα μέσα να διορθώσουμε προβλήματα που έχουν εντοπιστεί. Ωραία. Επανερχόμαστε στον εισηγητή μας, τον Κάρλ Σλόιτερ. Το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο δεν επιθυμεί το λόγο. Ναι, αλλά εμείς θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη του Συμβούλιο. Προς το παρόν δεν έχει διαμορφώσει γνώμη το Συμβούλιο. Πρόκειται για πρώτη ανταλλαγή απόψε, δικαιούται και το Συμβούλιο να επιφυλαχθεί και να επανέλθει σε μεταγενέστερη συνεδρίαση. Οπότε έχετε το λόγο κύριε Σιγητά για τις τελευταίες σας παρατηρήσεις για σήμερα. Και δώστε μας και μια, μερικές προτάσεις για το χρονοδιάγραμμα σε ό,τι φορά τη συνέχεια της συζήτησης. Μικρόφωνο. έκανα ένα σχόλιο στα γαλλικά προς τους φίλους της Βελγικής Προεδρίας. Φάνηκε από τη συζήτηση ότι η κατάσταση είναι εκεί και εμείς θέλουμε κάτι ψή. Κάθε χώρα λέει κάτι ότι μπορεί για τις διαπραγματεύσεις. Αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο, αλλά το ακόμη καλύτερο μπορεί να είναι μια κατάσταση με συνθήκες ίσου και θεμητού ανταγωνισμού με ένα πάγιο και ασφαλές νομικό πλαίσιο που ο καθένας θα ξέρει τι ισχύει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν ότι τους περάσει από το μυαλό γιατί ισχύει η συνθήκη. Αυτό έκαναν τα τελευταία 50 χρόνια. Γι' αυτό είχαμε και τόσο πολλές και διαφορετικές διαπραγματεύσεις. Είμαστε σε μια κατάσταση που δεν ικανοποιεί κανέναν δηλαδή σήμερα. Αλλά ο μόνος τρόπος για να ξεφύγουμε από αυτό είναι να αξιοποιήσουμε τη συνθήκη, γιατί αυτή, έχω, αυτή τη συνθήκη έχουν υπογράψει και εγκρίνει όλες οι χώρες, ακόμη και σε μερικούς δεν αρέσει. Οπότε θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να περάσουμε από την κατάσταση Α στην κατάσταση Β. Από μια κατάσταση που μας δυσαρεστεί σε μια που θα μας ικανοποιεί. Ο κύριος Κάσπαρη μίλησε για νομική ασφάλεια. Φυσικά, χρειαζόμαστε μια βεβαιότητα και νομική ασφάλεια. Γιατί η αστάθεια και η αβεβαιότητα δεν βοηθάει κανέναν. Θέλουμε λοιπόν μια μεταβατική περίοδο που θα λαμβάνει υπόψη αυτή την ανάγκη της νομικής ασφάλειας. Αλλά η παρούσα κατάσταση δημιουργεί έλλειψη νομικής ασφάλειας, γιατί θα πρέπει να δούμε ποιος προσδιορίζει τους κανόνες που ακολουθούν οι διάφορες εμπορικές συμφωνίες. Ακόμη και αν είχαμε μακροχρόνιες μεταβατικές περιόδους με πολλές εξαιρέσεις, ακόμη δεν θα αποκαθιστούσαμε μια νομική ασφάλεια. Ιδιαίτερα σε περίπτωση που ανακύψουν ε, συγκρούσεις και διαφορές. Τι δικαιοδοσία θα ισχύσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ποιος θα επιλαμβάνεται για να διευθυνθεί τις διαφορές. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένα είδος δημοκρατικού ελέγχου. Οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους κανόνες που θεσπίζει η συνθήκη και να βρούμε μια μεταβατική περίοδο που θα ορίσουμε τη διάρκεια της. Δεν απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη ρήτρα εκπνοής, ίσως μια άλλη φορά. Η κυρία Σαρνές, Δεσσαρνές, έθιξε παρόμοια ζητήματα με αυτά που επισήμανε ο κύριος ε, Κάσπαρη και Καντέρα Ρίφα, μάλλον θα είσαι ο σκιώδης δεν έχει οριστεί ακόμη, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα είσαι εσύ ο σκιώδης, οπότε θα συζητήσουμε σίγουρα μαζί. Εκτός μικροφώνου το σχόλιο του κυρίου Ντάρτμουτ. Προσπάθησα να διαχωρίσω τη δική σου θέση και των Γάλλων. Εν πάση περιπτώσει, ακόμη και αν η Σουηδία έχει τέτοιε εμπορικέ συμφωνίε, φαντάζομαι η Σουηδική κυβέρνηση θα προσπαθήσει, θα προτιμούσε να κρατήσει εκείνη την εξουσία, αλλά τώρα έχουμε νέα συνθήκη, νέους κανόνες και είμαστε και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να μην είστε με την κατάσταση αυτή, αλλά για άλλους είναι προτιμότερη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι είναι αδιανόητο. Ναι, αδιανόητο είναι οι νέε συμφωνίες να γίνονται ερήμην του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι αδιανόητο να παραμερίζεται πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην διαπραγμάτευση. Χαίρομαι πάντως που ήδη από τώρα ζητήσατε κατευθυντήριες γραμμές για το μέλλον της ε, επενδυτικής πολιτικής. Και φαντάζομαι θα το πραγματευτούμε αυτό σε επόμενες εκθέσεις. Καλό θα ήταν να διορθωθούν κάποιες ασυμβατότητες μεταξύ κάποιων στοιχείων των εμπορικών συμφωνιών και της συνθήκης και το θέμα της αποκατάστασης νομική ασφάλεια επίσης είναι πολύ σημαντικό. Και κάτι που ξέχασα προηγουμένω είναι η επενδύση χαρτοφυλακίου. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Αυτό το ερώτημα το θέτω για προβληματισμό γιατί ίσως το αναφέρω και στην έκθεσή μου. Ο κύριος Κάσπαρη μίλησε και για το χρόνο, την προθεσμία. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Καλύτερα να σπεύσουμε βραδέως και να προβλέψουμε όσο χρόνο χρειαζόμαστε για να καταλήξουμε σε μια σωστή πρόταση. Να μην φροντίσουμε πάση θυσία να επισπεύσουμε τα πράγματα, αλλά να, να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να ξέρουμε τη στιγμή της ψηφοφορίας τι ακριβώς θα ψηφίζουμε. Και φυσικά να ελέγξουμε όσο δυνατό περισσότερες συμφωνίες γίνεται. Ελπίζω και το Συμβούλιο να μας ενημερώσει κάποια στιγμή για το πώς εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο. Γιατί εκεί είναι που υπάρχουν τα εμπόδια στην αλλαγή. Γιατί αρχικά το Συμβούλιο ήταν αρμόδιο. Τώρα εκχώρησε κάποιες ε, αρμοδιότητες, αλλά πολλοί δυσανασχετούν με αυτή την εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Οπότε, ίσως μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου θα υπάρξουν προβλήματα παρά κοινοβουλίου, μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Αλλά θα πρέπει να συνεννοηθούμε για να δούμε πώ θα προχωρήσουμε γιατί μια τέτοια κατάσταση θα μας οδηγήσει σε έλλειψη νομική ασφάλεια αν δεν βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε. Αν δεν συμφωνήσουμε αυτό θα είναι το χειρότερο, είναι απευκταίο λοιπόν. όσοι είναι κατά της συμφωνίας θα προσπαθήσουν να καθυστερήσουν τη διαδικασία γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μπλοκάρει νέες συμφωνίες, να προσφύγει στα δικαστήρια για παλιές και το, το Κοινοβούλιο το ίδιο. Όλοι μπορούμε να κολλησιεργήσουμε, αλλά το θέμα είναι να γυρίσουμε τη σελίδα και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε καλύτερα στο μέλλον. Ξέρετε πόσο καιρό θα χρειαστείτε για τη σύνταξη της νομοδότησης. Θέλετε να κρατήσουμε τη συζήτησή σας παράλληλη με τη συζήτηση για τις εξωτερικές επενδύσεις. Περνάμε λοιπόν τώρα στο 14. για μια νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη. 2011-2020. οι συντονιστές τον Ιούλιο αποφάσισαν ότι θα γνωμοδοτήσουμε προς την αρμόδια επιτροπή την Ήτρε Προβλέπεται η υιοθέτηση της εκθέσεως στην Ήτρε στο τέλος Σεπτεμβρίου και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας και γι' αυτό η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η Δευτέρα Σεπτεμβρίου 12 μεσημβρινή. Λίγες μέρες έχουμε μπροστά μας. Ο Γιάνν Θαχαντήλ είναι ο εισηγητής μας, δεν μπορεί να είναι παρόν. Και θα δώσω το λόγο στο Στέντε. ο οποίος θα παρουσιάσει τη γνωμοθέτηση αυτή. Ζητά συγγνώμη ο κ. Ζάχαντελ. Μου έχει στείλει κάποια μικρά κείμενα τα οποία θα σας παρουσιάσω αλλάζοντας λίγο ε, την σύνταξη στην αγγλική γλώσσα. Λοιπόν, είναι σωστή η λογική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προχωρήσει στην ολοκλήρωση αυτής της νέας ενεργειακής στρατηγικής. Η στρατηγική αυτή από το 2011-2020 θα πρέπει να βασίζεται στην αηφορία, τον ανταγωνισμό, την διασφάλιση της προμήθειας και την αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουμε μαζί ε, τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Υπάρχει το θέμα της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας, των υποδομών, των τρόπων προμήθειας, των δικτύων προμήθειας. Όλα αυτά είναι κομβικά σημεία για τη διασφάλιση των προμηθειών ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Θα πρέπει να αναπτυχθούν λοιπόν συνέργειες στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες χώρες ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε τιμές της αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει με εμπορικές συμφωνίες να επιταχύνει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να προωθήσουμε το εμπόριο και στις νέες πηγές ενέργειας και στις νέες ενεργειακές τεχνολογίες. Ταυτόχρονα επιβεβαιώνουμε τον ρόλο που, έχει, που έχουν οι άμεσες ευρωπαϊκές επενδύσεις για τον εξοχρονισμό των υποδομών στις υποανάπτυξη χώρες. Μέσω ιδιωτικών και δημοσίων εταιρικών σχέσεων και κοινών προσπαθειών θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη συνεργασία μας με τις χώρες αυτές προς το αμοιβαίο συμφέρον και των όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω πώς ακριβώς φαίνεται στο γραπτό σας κείμενο, αλλά ζητάμε από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξουν την αλληλεγγύη στα πλαίσια της αντιμετώπισης των προβλημάτων και των προκλήσεων στην ενέργεια των 21ο αιώνα. Με βάση το άρθρο 194 ελπίζω ότι θα προχωρήσουμε με θετική ενέργεια. Ζητώ συγγνώμη για τον αποσπασματικό τρόπο που παρουσίασε τις θέσεις του κυρίου Ζαχραντήλ. Θα σημειώσω όποιες παρατηρήσεις κάνετε γύρω από το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έχουν το λόγο Ζαντό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Αυτό το οποίο με εκπλήσει είναι το ότι δεν βρίσκω στο σχέδιο αυτό τη συνένεση η οποία υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι στην Ευρώπη και στον τομέα της ε, ενέργειας και στον τομέα της στρατηγικής βασικός μας στόχος είναι η ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Το να βασίσουμε το σύνολο της προσπάθειας την οποία κάνουμε ε, στην διασφάλιση της προμήθειας της ενέργειας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι κάτι το οποίο θα χαρακτήριζα ανάποδο. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ενέργεια στην Ευρώπη μέσω των υποδομών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα δεν είναι μόνο ενεργειακό, είναι θέμα οικονομικό, είναι θέμα βιομηχανικό, είναι θέμα ανάπτυξης βιομηχανικών ικανοτήτων και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και στις εξωγωγικές αγορές. Ξέρετε ότι στην Κίνα έχουν επενδυθεί 230 δις σε τεχνολογίες οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον, 80 δις στις Ηνωμένε Πολιτείες και 25 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να εξοικονομήσουμε ενέργεια, να είμαστε ε, αποτελεσματικοί ενεργειακά και να εμείνουμε στη συνένεση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί στην πυρηνική ενέργεια δεν υπάρχει συνένεση και εκεί θα πρέπει να εμείνουμε και όχι να ανοίγουμε θέματα τα οποία δημιουργούν συζητήσεις και προβλήματα χωρίς τέλος. Νομίζω ότι η ιδέα μιας κοινή στρατηγικής για την ενέργεια θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε πέραν απλά της αναγνώρισης της αλληλεγγύης, της αρχής της αλληλεγγύης. Θα πρέπει να υπάρξουν ευρωπαϊκές επενδύσεις, αλλά το λεγόμενο ευρωπαϊκό μίξ θα εξαρτηθεί από όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν υποχρεώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ενέργειας και κάθε κράτος μέλος δεν θα πρέπει να αποφασίζει μόνο του, αλλά θα πρέπει και οι ευρωπαϊκοί κανόνες να τίθεται σε ισχύ. Ευχαριστώ κύριε Ζαντό. Έχετε τη δυνατότητα να καταθέσετε προτάσεις για να βελτιώσετε την πρόταση αυτή. Παρακολούθησα προσεκτικά αυτά που είπατε. Λοιπόν, δεν ξέρω, κάποιος άλλος συνάδελφος θα ήθελε το λόγο. Όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας ζητά συγγνώμη γιατί δεν είναι παρούσα. Διερωτώ με αν υπάρχει Γενική Διεύθυνση Εμπορίου που θέλει να πει κάτι. Όχι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στέρντι έχει ζητήσει το λόγο. Θα μεταφέρω το μήνυμα προς τον κύριο Ζαχράντιλ δεν έχει διευκρινιστεί η θέση μας για την πυρηνική ενέργεια. Ξέρω όμως ότι σε ορισμένες χώρες η πυρηνική ενέργεια κερδίζει θα έλεγα χώρο. Λοιπόν θα περάσω ό,τι άκουσα στον κύριο Ζαχράντιλ. Καλώς, ευχαριστώ. Το επόμενο θέμα είναι το τελευταίο στην ημερησία διάταξη πριν περάσουμε στη συνέντευξη των συντονιστών και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω τους συντονιστές να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση πέντε λεπτά μετά το τέλος της συζήτησης του επομένου θέματος. Συμφωνείτε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν το 15 είναι ανταλλαγή απόψεων για τις αγγιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η συγκητής μας μάλλον υπεύθυνη επιτροπή, αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμού και εμείς θα καταθέσουμε τη δική μας γνωμοδότηση. Ο Λόρδος Ντάθμορ είναι ο εισηγητής μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η γνωμοδότηση όταν συνταχθεί ουσιαστικά θα περιλαμβάνει ε, ενημερωμένες γνώμες. Τώρα θα περιοριστώ να υποβάλω μια όσο γίνεται σαφέστερη έκθεση του περιεχομένου. Προσθέτοντας ότι μπορεί να επαναλάβω λίγο αυτά που είπα πριν από έξι εβδομάδες. Πριν από έξι εβδομάδες έγιναν αυτά. Και αν έχει κανείς τόσο καλή μνήμη που να θυμάται τι είπα εγώ πριν από έξι εβδομάδες, ζητώ συγγνώμη για την επανάληψη. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους ε, ειδικού ε, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και της Κομισιόν με τους οποίους ε, συνεργάστηκα σήμερα το πρωί. Τους ευχαριστώ για το χρόνο τους, αλλά και για τη σαφήνεια των θέσεών τους. Περί τίνος πρόκειται ουσιαστικά. Υπάρχει μια εγγύηση που υπάρχει τώρα από τον προϋπολογισμό της, ε, της Ένωσης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 85 δις ευρώ για να... και θα πρέπει αυτό, αυτή η πρόβλεψη να ανανεωθεί τον Οκτώβριο του 2011. Πέραν αυτού υπάρχουν και άλλα δύο δις ευρώ εγγύηση που θα εγκριθούν ταυτόχρονα και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στα θεσμικά όργανα να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής των εργασιών τους. Πολύ λυπάμαι που δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή ο κύριος Σλάιτερ, γιατί ε, μεγάλο ε, μέρος των θεμάτων που ε, θέτει ε, δεν πρόκειται να καρποφορήσουν από ό,τι φαίνεται εδώ. Πρόκειται για έργα τα οποία, γιατί έχουμε πολλά προγράμματα για την κλιματική αλλαγή ήδη και την ανάπτυξη της υπαίθρου ε, τα ε, σχετικά δάνεια μπορούν και με τις συμφωνίες για τα δάνεια θα ανανεωθούν στην ε, Ιράκ, Καμπότζη, Ισλανδία, Λιβύη, Λευκορωσία θα καλυφθούν. Επίσης ο ρυθμός των χορήγησης των δανείων είναι καλός από την ΕΤΕΠ και τα μόνα επισφαλή δάνεια που είχαν ε, ήταν η Αργεντινή και η Ιουγκοσλαβία μετά από την πτώχευση. Η Αργεντινή ε, μέσα σε μία από τις πολλές οικονομικές κρίσεις και η ε, Ιουγκοσλαβία επειδή έπαψε να υφίσταται παρά το γεγονός ότι έγινε αναδιάρθρωση του δανείου στην Αργεντινή και δεν υπήρξε ηλική απώλεια. Το δάνειο στη Γιουγκοσλαβία ε, κατενεμήθη, επιμερίστηκε, επιμερίστηκε, καλύτερα να το πούμε, μεταξύ των δημοκρατιών διαδόχων του κράτους της Γιουγκοσλαβίας. Δεν θα τις αναφέρω, δεν θα τις απαριθμίσω όλες. Ιδιαίτερα γιατί οι Έλληνες συνάδελφοι έχουν πρόβλημα με ένα όνομα από μια πρώην Ιουγκοσταβική Δημοκρατία. Δεν υπήρξε λοιπόν απώλεια. Δεν υπήρχε, δεν ε, κατα... απώλεια. Να προσθέσω επίσης ότι η ΕΤΕΠ ε, έχει καλή κεφαλαιοποίηση, άρα μπορεί να δανείζει περισσότερα χρήματα χωρίς ε, να ε, χρειάζεται περισσότερο κεφάλαιο του επίπεδου 1. Επίσης, τα μεγάλα ποσά που ανέφερα είναι ανώτατα όρια, οροφές, δεν είναι στόχοι δηλαδή. Άρα προσδοκούμε ότι τα χρήματα που δίνονται, που δανείζονται με τα κριτήρια αυτά θα είναι σημαντικά λιγότερα ε, κατόγκων από το ποσό που αρχικά είχε προβλεφθεί μαζί με το, τα δύο δις ευρώ. Η τράπεζα θα προσπαθήσει να ε, πληρώσει στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη εμπορικούς και η πρόθεση είναι οι εγγύησει να καλύπτουν το πρόσθετο, τον πρόσθετο κίνδυνο ε, που αναλαμβάνει μέσα από αυτά τα μη εμπορικά δάνεια. Επίσης, να δούμε και το πρόσθετο ποσό που ζητήθηκε, που είναι ε, ένα συν 9 κατά 9%. Επίσης, κάτι που είπα και θα το αναφέρω περιληπτικά είναι ότι υπάρχουν σημαντικές πιέσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε η ΕΤΕΠ να δίδει περισσότερα αναπτυξιακά δάνεια και θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά τα αναπτυξιακά δάνεια ε, είναι πολύ εντατικά από άποψη διοίκηση και προσωπικού και απαιτείται περισσότερο προσωπικό, περισσότερη πρόσβαση ε, προς χορηγήσεις ούτως ώστε να συμπληρώνονται τα δάνεια και Αυτό είναι μια πρόσθετη λειτουργία, χωριστή πέρα από τις λειτουργίες ε, τις σημερινές της ΕΤΕΠ. Αυτό θα ήταν δυσανάλογα ακριβό εγχείρημα και ίσως καλό είναι οι συνάδελφοι να το έχουν υπόψη τους όταν επιμένουν να ζητούν η ΕΤΕΠ να ασχοληθεί περισσότερο με τα αναπτυξιακά δάνεια. Και σε αυτό το σημείο ε, ολοκληρώνω την εισαγωγή μου για να αρχίσουμε τη συζήτηση. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ας αρχίσουμε λοιπόν τη συζήτηση. Ο Ζορς Κούτας. Uh, uh, είναι σαφές ότι τα δάνεια τα οποία έχει χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αντιπροσωπεύουν περίπου τις μισές επενδύσεις τις οποίες έχει χορηγήσει η Παγκόσμια Τράπεζα. Είναι λοιπόν σημαντική η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και μπορεί να βοηθήσει κάποια προγράμματα που έχουν σαν στόχο τις κλιματικές αλλαγές, τις περιβαλλοντικές υποδομές, την προώθηση των αηφόρων μορφών μεταφορών, όπως επίσης και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν οι μικρομεσαίες, γιατί έτσι θα βοηθηθεί η οικονομική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα μπορούμε να ενισχύσουμε τις εταιρικές σχέσεις ανάμεσα στις χώρες της Ένωσης και αυτές τις χώρες και να καταπολεμήσουμε την φτώχεια που υπάρχει στις χώρες αυτές. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη παρατήρηση, ίσως όμως να έχει κάποια σημασία. Νομίζω ότι οι αιτήσιε αξιολογήσεις της αποτελεσματικότητας των δανείων είναι απαραίτητες. Διασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια, μειώνουν τα διοικητικά εμπόδια και νομίζω ότι εν πάση περιπτώσει τα μέσα τα οποία έχουμε ε, στην διάθεσή μας θα πρέπει να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήδη στην προηγούμενη συζήτηση είχαμε αναφερθεί στο σημείο αυτό. Το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει αναλάβει εντολή για το κλίμα, εκ πρώτης όψεως δεν μας δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και δυσκολίες, Υπό τον όρο όμως θα συμφωνήσουμε για τα κριτήρια χρηματοδότησης της ΕΤΕ και τα εχέγγυα εγγύησης που θα προταθούν. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοια κριτήρια για το τι σχέδια θα εξυπηρετούν αυτό το στόχο της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. Φαίνεται ότι το θέμα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, τα μεγάλα φράγματα, τα βιοκαύσιμα είναι πιθανά σχέδια και δεν αποκλείονται από την εντολή αυτή της ΕΤΕ. Γιατί να μην έχουμε μια τέτοια εντολή για τις κλιματικές αλλαγές. Τα σχέδια όμως που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις κλιματικές αλλαγές, τα μεγάλα φράγματα, το θέμα δέσμευσης άνθρακα, δεν εξυπηρετούν αυτόν τον αγώνα κατά των κλιματικών αλλαγών, θα πρέπει να αποκλείονται από την εντολή αυτή τη ΕΤΕ, κάτι που δεν ισχύει τώρα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Υπάρχει εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Στέφαν Άπερ. Χωρίς μικρόφωνο. draw the microphone closer to you, please. Παρακαλώ, να μιλάτε πιο κοντά στο μικρόφωνο, δεν σας ακούμε. Does this work? Ah, okay. okay. No, thank you very much. Uh, I don't... Ευχαριστώ. Δεν έχω να προσθέσω και πολλά. Πολύ εύγλωτα ο εισηγητής εξήγησε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι που απαιτεί ισχύουσα νομική βάση. Πάντως η διάταξη αυτή προβλέπει τον Οκτώβριο του 2011 ως καταληκτική προθεσμία. Οπότε αν δεν ληφθεί νέα απόφαση, δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ε, οι εγγυήσει του κοινοτικού προπολογισμού, γιατί υπάρχει αυτή η ρήτρα εκπνοή. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο για να σα εξηγήσει τα των κλιματικών αλλαγών. That's all right. Thank you, Mr. Chairman. Δεν έχω να προσθέσω πολλά. Θα ήθελα να επισημάνω πάντως το πιο σημαντικό σημείο που είναι ότι η ΕΤΕ σε τέτοιου είδους εξοκοινωτικές δραστηριότητες ε, εργάζεται με βάση πολιτικές εντολές. Αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι να εφαρμόζουμε τις κοινοτικέ πολιτικές. Και αυτό είναι το σημείο αφετηρίας. Τώρα, ως προ το, στο κριτήριο για τι κλιματικέ αλλαγέ και τι ασυναφεί επενδύσει. Φυσικά είμαστε πρόθυμοι να παρουσιάσουμε τα κριτήρια και τον ορισμό των προγραμμάτων προκειμένου να συμπεριληφθούν στην εντολή για την κλιματική δράση. Αυτό είναι προφανές γιατί δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Το σημειώνουμε πάντως και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Πάντως πιστεύω ότι δεν είναι η τράπεζα αυτή που αποφασίζει, αλλά εσείς, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Γιατί δεν υπάρχει μόνο μια κοινοτική πολιτική, υπάρχει και η πολιτική ενεργειακής ασφάλειας και η ε, πολιτική κλιματικής δράσης. Οπότε αν χρηματοδότηση γίνεται μόνο ε, υπό το κεφάλαιο της ενεργειακής ασφάλειας, δεν εμπίπτουν στο στο... στην εντολή των 2 δισεκατομμύριων για τις κλιματικές αλλαγές. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς. Να παρουσιάσουμε τα κριτήρια, να είμαστε διαφανείς, να συμμορφωθούμε με τις δικές σας προϋποθέσεις και απαιτήσεις και να αποφασίσουμε ότι αποφασίζεται στο κατάλληλο επίπεδο. Ευχαριστώ και ολοκληρώσαμε και το σημείο αυτό. Ο εισηγητής, ο κύριος Στάρτμουντ, θα ήθελα να πω απλώς ότι πριν από έξι εβδομάδες είχα πει ότι η ΕΤΕ δεν ήταν ούτε μισή παγκόσμια τράπεζα. Βέβαια το μέγεθος είναι το πάνω, αλλά το θέμα είναι ότι η ΕΤΕ ε, πραγματοποιεί πολύ σημαντικές δραστηριότητες και οι δράσεις της έχουν σημαντικά αποτελέσματα και συνέπειες. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ότι σπάνια συμφωνώ με τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, αλλά αυτή τη φορά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ότι είναι πολύ σημαντικό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να λαμβάνουν σημαντικό και μερίδιο των επιδοτήσεων. Ή μάλλον θα το πω με άλλα λόγια, ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί πλήρης πρόσβαση των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα δάνεια της ΕΤΕ. Και αυτό θα το προσθέσω στη γνωμοδότησή μου. Η ΕΤΕ θα έχει εντολή και για τις κλιματικές αλλαγές. Και φυσικά αυτή η εντολή θα πρέπει να προσδιοριστεί. Το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει το εύρος αυτής της εντολής. Δεν ξέρω ποια θα είναι η έκβαση των συζητήσεων. Τώρα, αυτή τη φορά το σχόλιο για την ενεργειακή ασφάλεια. Με κλώνησε κάπως, γιατί είναι και εύλογο και ευκταίο. Ορισμένα δανεία έχουν μη εμπορικό στόχο και πρόθεση εξασφάλισης του ενεργειακού ανεφοδιασμού. περιμένουμε με ανυπομονησία την επόμενη φάση της συζήτησης, ε, τότε θα έχουμε και το έγγραφο. Καλώς. Ολοκληρώνεται και αυτό το σημείο. Να σας υπενθυμίσω ότι το σχέδιο γνωμοδότησης θα συζητηθεί στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου. Διάφορα. Δεν έχουμε διάφορα. Οπότε σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία σας. Η επόμενη μας συνεδρίαση θα γίνει στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου. Σε 9 το πρωί θα αρχίσουμε στις 28 Σεπτεμβρίου. Σε 5 λεπτά θα συνεδριάσουν οι συντονιστές. Οι υπόλοιποι παρακαλώ να εγκαταλείψουν την αίθουσα. There's another...